Και περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη αυτή τη Συνόδου. Για την ημερήσια διάταξη καταρχήν έχω ένα αίτημα του κυρίου συναδέλφου Φαντάλε που γραπτός μου γνωστοποίησε ότι για την ημερήσια διάταξη θα ήθελε να παρέμβει. Παρακαλώ κύριε Φαντάλε μπορείτε να παρέμβετε, έχετε τον λόγο. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, dit weekend is bekend geworden dat uh, de heer Van Rompuy aan Egypte voor 5 miljard aan steun heeft toegezegd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 daarom graag op korte termijn een uitleg van van rompuy plus een debat en ik wil u vragen die vraag mee te nemen. wanneer kunnen wij daarover debatteren? mogelijk in februari al? Ίσως θα ήταν ο Φεβρουάριος ένας καλός χρόνος για να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Φαντρομπέ. Είναι σημαντικό να το συζητήσουμε. Δεν είναι θέμα το οποίο αφορά τι εργασίε αυτή τη Συνόδου. Θα ήμουν ευγνώμων αν ε, διαβιβαστεί αυτό το αίτημα, θα διαβιβαστεί στου αρμόδιου στην αρμόδια αρχή και θα διευκρινιστεί με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να διαβουλευτούμε επ' αυτού του θέματο. Καταρχήν για διαδικαστικό ζήτησε τον λόγο ο κύριος Λάιχτφριντ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όχι για την ημερήσια διάταξη, αλλά για τις προηγούμενες τοποθετήσεις σας. Μια σύντομη ανακοίνωση. Πριν από κάποιο καιρό υπήρξε η εξή κατάσταση. Ε, από τρεις συναδέλφους αυτού του σώματος υπήρξε η υποψία νομοθεσία μέσω πληρωμών να ε, ασκηθεί και ο αρμόδιος ε, ε, αυστριακός συνάδελφος ο οποίος ε, παρετήθηκε προσήχθη στα δικαστήρια και καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση ιδιαίτερα με το αιτιολογικό ότι με κάποιον ευρωβουλευτή, δεν πρόκειται για κάποιο μικρό δήμαρχο, αλλά για κάποιον συνομοθέτη στο υψηλότερο επίπεδο της νομοθετικής εργασίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αυτή ήταν η ανακοίνωσή μου. Θα ήταν ίσως ε, να διαβιβαστεί αυτό το θέμα και στο ε, Συνταγματικό Δικαστήριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προς ενημέρωση. Ο κύριος Τάνοκ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικό. Η πολιτική μου ομάδα έχει υποβάλει ένα αίτημα σήμερα το απόγευμα προκειμένου να γίνει μια συζήτηση την Τρίτη παρουσία της ε, ΥΠΑ της εκπροσώπου ε, για το Μαλί. Έχουμε μια στρατηγική επέμβαση από ένα κράτος μέλος με την υποστήριξη της δικής μου της χώρας απορρίφθηκε και τεχνικού λόγου. Δεν καταφέραμε να υποβάλουμε το αίτημα μέχρι τι 4 το απόγευμα. Επομένω, θα ήθελα να σα ζητήσω να ψηφίσει η Ολομέλεια προκειμένου να καταφέρουμε να εντάξουμε το σημείο αυτό στη μερίσια διάταξη. Πολύ σημαντικό το σημείο αυτό για την ομάδα μου. Ευχαριστώ. Ε, λυπούμε Προφανώς αυτό το αίτημα δεν διαβιβάστηκε και δεν το έχουμε ενώπιόν μας. Ηρεμήστε παρακαλώ κύριε Ποντή. Κύριε Οντή, δεν ε, διαβιβάστηκε επισήμω το έτοιμά σα. Θα δούμε γιατί δεν συνέβη αυτό. σω και εσεί μπορείτε να διακριβώσετε στην ομάδα σα τι συνέβη. Δεν έχουμε κάποιο επίσημο τέτοιο αίτημα μέχρι τι 4 η ώρα, 16.00 σήμερα το απόγευμα, για να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη. Λυπούμε. Ο κύριο Ντονζόν, παρακαλώ. Oui, Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά θεωρώ λυπηρό το ότι για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, δηλαδή μια ένοπλη σύραξη που ξέσπασε και η οποία αφορά ένα κράτος μέλος, το οποίο έχει μάλιστα υποστεί και απώλειες στο Σαββατοκύριακο και αφορά μια περιοχή για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν κρίνει μια στρατηγική εδώ και περίπου δύο χρόνια Θέλω να την υπενθυμίσω τη στρατηγική αυτή και εμείς έχουμε ζητήσει από τις επιτροπές εδώ στο Κοινοβούλιο να εφαρμοστεί στην πράξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα είναι έτοιμη να ξεκινήσει στη χώρα αυτή ε, μια αποστολή, ε, στο Μαλί συγκεκριμένα, και λυπούμε γιατί δεν έχουμε ένα συνομιλητή. Πέντε ώρες την Τετάρτη θα ασχοληθούμε με την κοινή πολιτική ε, ασφάλειας και άμυνας και την κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν μπορούμε να βρούμε χρόνο για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Είναι λυπηρό και για εμάς και για το πολύ θλιβερό θέαμα το οποίο παρουσιάζουμε στους συμπολίτες μας. Παρακαλώ κύριε Θέλω μόνο για αυτές τις αναφορές να πω ότι δυστυχώς από καμιά ομάδα δεν ζητήθηκε αυτή η συζήτηση να διεξαχθεί. Όμως το θεωρώ απόλυτα αναγκαίο να γίνει αυτό. Και θα πίστευα, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να ζητηθεί από την κυρία Άστον η περίοδο συνόδου να είναι αφορμή να προσέλθει η κυρία Άστον στην Ολομέλειά μα. Επί αρκετό χρονικό διάστημα δεν έχει προσέλθει. Είναι πολύ σημαντικό να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση. Παρακαλώ, διαβιβάστε αυτή την παράκληση προ την κυρία Άστον. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Χάρμ για την γενική σύγχυση δεν ξέρω αν πρέπει να την επαυξήσω αλλά σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες η κάθε Άστον πρότεινε όχι την Τετάρτη αλλά την Τρίτη, δηλαδή αύριο να προσέλθει στο Στρασβούργο σε εμά. Και πρότεινε επίσης με εμά αν θέλουμε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη, να συζητήσει και για το Μάλι και για τη Συρία, αλλά και για το αίτημα το οποίο εξεφράστη σε σχέση με τη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο. Εγώ εξ ονόματο ομάδα μου μπορώ να πω ότι είμαστε υπέρ να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη και να μπορέσει να έρθει η κυρία Άστον εδώ αύριο και να συζητήσουμε αυτά τα τρία θέματα μαζί της αύριο εδώ. Ευχαριστώ. Δεν επαυξήσατε τη σύγχυση κυρία Χάρμς, αλλά μάλλον ε, αποσαφηνίσατε κάποια πράγματα. Η κυρία Άστον δεν, είχε επαφή, δεν ήρθε σε επαφή μαζί μου αυτό το Σαββατοκύριακο και πρέπει να το διαπιστώσω και να το πω αυτό, ώστε κάποιες φήμες που υπάρχουν να διαλυθούν. Ωστόσο, είχα τηλεφώνημα από τις υπηρεσίες του σώματος το Σαββατοκύριακο ότι το γραφείο αυτής της, κυρία κυρίας Άστον υπέβαλε αυτό το αίτημα με την επισήμαση ότι δεν θα, μπορούσε το, δεν θα γινόταν το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με την συνθήκη να προσέλθει στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπως ήταν υποχρεωμένη και να προσέλθει και το Νοέμβριο στην Ολομέλεια. Στη συνέχεια αμέσω ε, ζήτησα από το γραφείο μου να έρθει σε διαβουλεύσει με τι κοινοβουλευτικέ ομάδε. Αν επιθυμούν οι κοινοβουλευτικέ ομάδε του Κοινοβουλίου αλλαγή τη ημερήσια διάταξη. Διότι είναι προπόθεση βασική αυτό. Σήμερα μέχρι τι 16.00 πρέπει να έχουμε τα αντίστοιχα αιτήματα για αλλαγέ ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξή μα. Καμία ομάδα δεν το ζήτησε αυτό. Καμία ομάδα δεν ετήθηκε αλλαγή τη ημερήσια διάταξη. Όχι, όχι. Δεν είναι κυρίαρχο το Κοινοβούλιο να αποφασίζει κατ' Έχουμε κανονισμό και πρέπει να τον τηρούμε. Λυπούμε. Τότε η ομάδα σας μέχρι τις 16.00 έπρεπε να είχε θέσει το θέμα. Κύριε Ντέιβις, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση και κρίνοντα από την γενικότερη ατμόσφαιρα στην αίθουσα ότι οτιδήποτε και να λέει ο κανονισμό, εσεί πρέπει να αποφασίσετε. Και σίγουρα πάρα πολλοί εδώ θέλουμε να ενταχθεί το ζήτημα του Μάλι στην ημερήσια διάταξη τη Ολομέλεια. Επομένω, κύριε Πρόεδρε, δική σα την εκκρατική ευκαιρία. μην κρύβεστε πίσω από τον κανονισμό. Oh, Λοιπόν, κύριε Τέβη, τέλειο όταν εσείς λαμβάνετε απόφαση επί θέματος αρχής ε, ότι η ελαστικότητα αυτή πρέπει να εφαρμόζεται αντίθετα με την απόφαση του Προέδρου να τηρηθεί ο κανονισμός. Τέλειο αυτό, διότι διαφορετικά ασκούνται πάντα επικρίσεις ότι δεν, ασκώ, δεν τηρώ εγώ τον κανονισμό. Τώρα, ότι εσεί μου ζητάτε αυτό, ευχαριστώ για την επισήμαση. Θα το κάνω ευχαριστώ. Σα λέω λοιπόν τι προβλέπει και τι λέει ο κανονισμό. Είναι σαφέστατο ο κανονισμός. Η μερίσια διάταξη μετά από την έγκρισή τη, εκτό σε σχέση με το άρθρο 142 ή μετά από πρόταση του Προέδρου δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή θα μπορούσα εγώ να ζητήσω να αλλάξει η μερίσια διάταξη. Εντάξει, καλώς, έστω. Κυρία Χάμς, Έχω κατανοήσει το αίτημά σας, μη φοβόσαστε, το κατάλαβα πολύ καλά. Προσπαθώ μόνο, χωρίς να παραβιαστεί ο κανονισμός, να ανταποκριθώ στο αίτημά σας, στις επιθυμίες σας. Η συζήτηση θα γίνει την Τετάρτη. Η κυρία Άστον όμως είπε ότι μπορεί να προσέθει μόνο την Τρίτη. Λοιπόν, καταρχήν θα προσπαθήσω να γνωστοποιήσω στην κυρία Άστον καταρχήν ότι επιθυμείτε να προσέλθει σε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή τι, την Τετάρτη. Αν την Τετάρτη όμως δεν μπορεί, αν την Τετάρτη δεν μπορεί, τότε με του Προέδρου των Κοινοβουλευτικών Ομάδων θα κάνω την προσπάθεια το πρόβλημα αυτό να το επιλύσω μέχρι αύριο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο σήμερα, αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνουμε, η συζήτηση προβλέπεται για την Τετάρτη. Θα προσπαθήσω για την Τετάρτη να έχουμε την κυρία Άστον εδώ, η Λέδη Άστον. Αν όμω δεν μπορεί να προσέλθει την Τετάρτη με κανένα τρόπο, θα συζητήσω με του Προέδρου των Κοινοβουλευτικών Ομάδων πώ μπορούμε να διαξαγάμε αυτή τη συζήτηση, υπό ποιε προποθέσει. Όμω, διαπιστώνω κυρίε και κύριοι ότι εγκρίνατε ότι σε περίπτωση αμφιβολίας για την ερμηνεία άρθρων του κανονισμού για την ημερήσια διάταξη θα αποφασίζει ο πρόεδρος. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Όχι, δεν είναι άπαξ αυτό, είναι θέμα αρχή. Θα μπορεί να γίνεται έτσι. Αυτό θα καταχωρηθεί και στα πρακτικά ω παρατήρηση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, κύριε Άντορ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, πρώτα απ' όλα καλή χρονιά σε όλους. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική μια πληροφορία που πρέπει να σας πούμε ότι η Αντιπρόεδρος Άστον είναι διαθέσιμη αύριο να συζητήσει το θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο αν ενδιαφέρεστε. Δυστυχώς δεν μπορεί την Τετάρτη. Γιατί λόγω της, ε, του προγράμματος που έχει. Ήθελα απλά να σας το γνωστοποιήσω. Πρόεδρος. Λοιπόν κύριε Άντορ, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Άντορ, σας ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε φτάσει ως εκεί και το είχαμε διαπιστώσει αυτό το οποίο μας αναφέρατε εσείς. Λοιπόν, με την κάθε άστον θα συζητήσω αυτό το θέμα. Όμως από πλευράς αρχής διαπιστώνω και λέγω, αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Συμβούλιο, εντάξει. Σε κανένα εθνικό κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε κάποιος υπουργός, γυναίκα ή άνδρα, άνδρας, να μην ακολουθήσει αίτημα του κοινοβουλίου και να μην προσέλθει. Und ich stelle nun και διαπιστώνω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απίφθινε αυτό το αίτημα κατεπηγόντως ε, να προσέλθει η ύπατος εκπρόσωπος την Τετάρτη στην Ολομέλεια. Λοιπόν, αυτό θα το συζητήσω καταρχήν μαζί της. Αν υπάρχουν κατεπήγοντες λόγοι που δεν μπορούν να αποφευθούν, θα, μπορέσουμε να, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιο συμβασμό για να επιληθεί το πρόβλημα. Αλλά το θέμα αρχής είναι, και πρέπει εδώ να διαφωνήσω, δεν μπορεί κανείς ως μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ω μέλος του Συμβουλίου ή ε, ύπατο εκπρόσωπο να πει Δεν θα πάω εγώ στην Ολομέλεια γιατί δεν μου το επιτρέπει η μερίσια διάταξη που έχω και οι αντιλημμένε μου υποχρεώσει. μια τέτοια πράξη ασέβεια δεν μπορεί να δεχθεί το Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, και περνάμε στη σημερινή ημέρα. Δεν έχουμε κάποια αιτήματα για αλλαγέ από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη για την περίοδο Συνόδου. Περνάμε στην πέμπτη τώρα. Για την πέμπτη. Για την πέμπτη η κοινοβουλευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς ζήτησε να υπάρξει μια τροποποίηση των κατεπηγόντων. Έχει τον λόγο η κυρία Τσίμερ για αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προηγούμενα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό δηλώσατε κάτι σε σχέση με την δολοφονία των τριών γυναικών, Κούρδων γυναικών ακτιβιστριών στο Παρίσι. Είμαστε γνώμονες γι' αυτό και τουλάχιστον είναι κάτι το ε, ξεχωριστό, απόλυτα ξεχωριστό και μοναδικό στην Ευρώπη να δολοφονούνται με τέτοιο τρόπο άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θέλω να ζητήσω εξ ονόματος της ε, ομάδας μας να πάμε ένα βήμα παραπέρα και την Πέμπτη υπό τα κατεπήγοντα το θέμα για τον Μπαχρέιν στην ημερήσια διάταξη να το αντικαταστήσουμε με ένα σημείο της ημερήσια διάταξη που θα αφορά τη δολοφονία των τριών ακτιβιστριών ε, Κούρδων γυναικών στο Παρίσι και να έχουμε και ένα σύντομο πρώτα, ε, κείμενο πρόταση ψηφίσματο που θα εγκριθεί, θα τεθεί σε ψηφοφορία προς έγκριση. Θα ασχολείται αυτό το ψήφισμα με, φυσικά με το ότι καταδικάζουμε στεναρά αυτή τη δολοφονία. Δεύτερον, ότι παρακαλούμε τι ε, γαλλικέ αρχέ και ζητούμε από αυτέ να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι του για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Και τρίτον, η διαδικασία διαβουλεύσεων και συζητήσεων μεταξύ τη τουρκική κυβέρνηση και του Ετζαλάν να υποστηριχθεί. Την υποστηρίζουμε εμεί αυτή τη διαβούλευση. Αυτό είναι το αίτημα τη ομάδα μα. Ευχαριστώ. Κυρία Τσίμερ, να σα ρωτήσω, λέει ο πρόεδρο, είχα ζητήσει το σημείο αυτό να αντικαταστήσει το θέμα του Μπαχρέν στην ημερήσια διάταξη και το προσθέτουμε αυτό. Θέλει κάποιο να λάβει τον λόγο υπέρ του αιτήματο τη κυρία Τσίμερ, παρακαλώ. Κάποιο θέλει να λάβει τον λόγο εναντίον. Κύριε Τάνοκ, υπέρ ή κατά. Okay. Okay. Exceptionally. Okay. Ε, Πολύ καλά. Είναι κάποιο ο οποίο θέλει να λάβει τον λόγο εναντίον εφόσον είσαστε εσεί υπέρ. Κύριε Σβόμποντα, εσεί είναι πραγματικά στη γερή δολοφονία και την καταδικάζουμε. Μόνο την καταδικάσουμε μπορούμε. Και φυσικά είναι σαφέ ότι οι γαλλικέ αρχέ θα πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι του να διαλευκανθεί η υπόθεση. Θα το προτιμούσα όμω αν θα είχαμε μια δήλωση Επιτροπή και Συμβουλίου στην επόμενη συζήτηση κατά την περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου, όταν θα γνωρίζουμε και περισσότερα. Ελπίζουμε για τη διαδικασία ειρήνευση ε, μεταξύ των, για τι διαβουλεύσει δηλαδή μεταξύ τουρκική κυβέρνηση ε, και Κούρδων. Αυτό θα ήταν πιο σοβαρό αν τότε το συζητούσαμε και γι' αυτό αν συμφωνείτε, τουλάχιστον εγώ θα ήθελα να θέσω το αίτημα να μην συζητήσουμε σε αυτή την περίοδο συνόδου, αλλά την επόμενη περίοδο συνόδου. Και έτσι να έχουμε και το θέμα τη ε, ειρηνευτική διαδικασία και της δολοφονίας που θα ενταχθούν σε ένα θέμα από κοινού. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, να σα ρωτήσω λοιπόν, δέχεστε αυτό το αίτημα, αυτή την τοποθέτηση. Εντάξει, ωραία λοιπόν. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν εσείς ως κοινοβουλευτική ομάδα θέτατε αυτό το θέμα, ε, μπορούσατε να θέσετε αυτό το θέμα για την επόμενη περίοδο συνόδου. Παραμένει λοιπόν χωρί ε, αλλαγέ, η ημερήσια διάταξη